σωστά αγγλικά να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Για την έκθεση του κ. Γκουαλτιέρη για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρώτη ψηφοφορία, μία ενιαία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας. The vote is closed. ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία για σήμερα. Έκθεση Swinburne για τις εξουσίες της κυρίας Swinburne, διορθώνει πρόεδρος, για τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή κυρώσεων. Πρώτα θα ψηφίσουμε τροπολογία 2 5 και 8 14 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Πέρας ε, ψηφορίας εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχος. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφές το αποτέλεσμα, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Εντάξει, λέει η Πρόεδρος, να το ελέγξουμε, μια και και πρώτη φορά που προεδρεύω για ψηφοφορίες. Στο δεύτερο τμήμα, λοιπόν, της τροπολογίας υπαριθμών 1. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ έναρξη της ψηφοφορίας. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 1. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 λοιπόν τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Σαφώς. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία περιθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε αυτό αν θα θέλατε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 7. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία της προτάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται το, η ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ονομαστική κλίση. Έναρξη τη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Το τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη για τις ψηφοφορίες. Πρόκειται για την ε, έκθεση και τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Λίμα του Περού. Να ξεκινήσουμε την παράγραφο 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. And I close the electronic vote. Πέρας. Εγκρίνεται. Okay. Then we come to amendment 1. Who is in favor? Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της ε, παραγράφου 14 τμήμα πρώτο. Πέρας εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε και πάλι άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική πέρασε εγκρίθηκε παράγραφος 16 τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Παράγραφος 10, όχι, μη συγχωρείτε, απορρίφθηκε. Άρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος 24, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίθηκε. Παράγραφος 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 29. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Παράγραφος 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 33 τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Παράγραφος 35 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επίσης εγκρίθηκε και τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Παράγραφος 36, τροπολογία 10, υπέρ. Κατά, αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ. Α, συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Απλώς άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με μεγάλη πλειοψηφία. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο, παράγραφος 39, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Με συγχωρείτε. Λάψους. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίθηκε παράγραφος 43 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με σαφή πλειοψηφία 51 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 55, τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 56, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 60 τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 11 υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές Φαίνεται ότι πέρασε, αλλά θέλω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχει εγκριθεί. Αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ. Με συγχωρείτε, I ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, X υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε αυτή την αιτιολογική σκέψη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ηλεκτρονικής εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την πρόταση στο σύνολό της υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στις ε, αιτιολογήσεις ψήφου. Θα ήθελα οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν να αποχωρήσουν για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε οι υπόλοιποι.